Η συγγήτρια είναι η κυρία Μούτζη. Να περάσουμε στην ψηφοφορία. Ε, συμβαστική 1 υπέρ, παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ, παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 8 καταπίπτει. Η 11 υπέρ. Κατά εποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θα ψηφίσουμε μόνο το δεύτερο τμήμα της 10 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές απορρίπτεται. 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφής η κατάσταση οπότε να κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση άρχεται Α, δεν λειτουργεί το μηχάνημά σας. Και τι ψηφίζετε παρακαλώ. Μάλιστα. Λοιπόν, παρακαλώ να επαναλάβουμε την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. την τροπολογία 11, με συγχωρείτε που την ξέχασα. Την 11 λοιπόν ψηφίζουμε υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ωραία. Συμβαστική 2 υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές Λοιπόν, ηλεκτρονικός έλεγχος για την συμβαστική 2 άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίνεται. Τροπολογία 23 υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 24 υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ με την προφορική τροπολόγηση που έχει το κείμενο 28 λοιπόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συγγνώμη 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονική παρακαλώ, άρχεται. Εγκρίνεται 18 υπέρ 4 κατά. Και συγχαίρουμε την εισηγήτρια. βαλε Ωραία, οπότε στις 10 και μισή, δηλαδή σε 5 λεπτά, σε 5 λεπτά λοιπόν, θα έχουμε την κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Απασχόλησης για να ασχοληθούμε με το θέμα της κατάστασης στην αγορά εργασία που ευνοεί το εργασίας που ευνοεί το συνδυασμό